να κοιτάξουμε το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης, να την εγκρίνουμε αν θέλετε, αν συμφωνείτε. Και περνάμε τώρα στην έγκριση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης. Έχετε καμία ερώτηση, εγκρίνετε τα πρακτικά. Ωραία, σας ευχαριστώ. Μετά έχουμε να κοιτάξουμε την έκθεση Λιμπράτσκι. Δεν είναι όμω εδώ ο κύριος Λιμπράτσκι και γι' αυτό θα περάσουμε στη δική μου έκθεση για τις ε, στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων. Θα ήθελα να αναφέρω στην Επιτροπή το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου της 30ης Ιουλίου. Το βασικό πρόβλημα το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται είναι το παράδειγμα 1, όπου το Συμβούλιο επιμένει στη συναπόφαση, ενώ η Επιτροπή θα ήθελε να υπάρχουν ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Ούτε η Πολωνική Προεδρία, ούτε η Επιτροπή έχουν λάβει εντολή να επαναχωρήσουν σε σχέση με τις θέσεις αυτές, άρα προσπαθώ να βρω μια συμβαστική λύση και με τους δύο σε ό,τι αφορά τις ε, τροπολογίες της Επιτροπής μας για τις, τα όρια εκπομπών ε, Ευρωπαϊκή Επίπεδου και τους ταχογράφους, συμφωνήθηκε να συνεργαστούμε και να καταθέσουμε ενδεχομένω νομοθετικές προτάσεις. Το Συμβούλιο αποδέχτηκε τις τροπολογίες της Επιτροπής μας για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων και αποδεχθήκαμε το αίτημα της Μάλτας για απόκληση από τα όρια αυτά. Αυτή η εξαίρεση δικαιολογείται λόγω γεωγραφικής θέσης και είναι περιορισμένη στη φύση της. Και όταν ο αριθμός οχημάτων που έχουν καταχωριστεί στη Μάλτα έχουν φτάσει τα 100, ο κανονισμός θα ισχύσει και για τη Μάλτα. Ο επόμενος τρομερής διάλογος κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει χώρα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Δεν έχω ακόμα στην διάθεσή μου ακριβή ημερομηνία. Θα σας ενημερώσω. Και σκοπός μου είναι να προσπαθήσω να πετύχω συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. σε ό,τι αφορά την έκθεση Simpson για τις μεταφορές εμπορευμάτων οδικός και ό,τι αφορά τις στατιστικές καταγραφές. Η κυρία Μάισνερ ζήτησε το λόγο. Okay. Yeah, uh, Thank you very much, Chair. I don't have... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, γιατί πραγματικά πρόκειται για διατύπωση και νομίζω ότι ο πρόεδρος ανέφερε όλα τα ότι Είναι σαφή τα πράγματα με τη Μάλτα, αν είναι διαφορετικές οι συνθήκες που επικρατούν σε ό,τι αφορά τις μεταφορές στη Μάλτα, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για απόκληση. Άρα δικαίω και ζητήθηκε. Και συμφωνώ και σε όλα τα υπόλοιπα με αυτά που είπε ο Πρόεδρος. Θα ξαναμιληθούμε για ένα τελικό τριμερή διάλογο και ελπίζω γοργά να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για άλλη μια φορά για την έκθεση. Νομίζω ότι η πρόταση τώρα σε ό,τι αφορά τη διατύπωση if appropriate που χρησιμοποιείται συνήθως από την ε, Επιτροπή σε ό,τι αφορά το Euroclass και Στην κάλυψη από ταχογράφους. Θεωρώ ότι είναι κάπως αδύναμη η διατύπωση. Θα ήθελα το as soon as possible να συμπεριληφθεί, το ταχύτερο δυνατόν, γιατί ο βασικός στόχος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση των εκπομπών. Και αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί και στην πράξη, να μην παραμείνει στη θεωρία. Άρα, θεωρώ ότι η διατύπωση θα πρέπει να είναι λίγο πιο έντονη προκειμένου να υπάρχει και αποτέλεσμα. Κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και δεν ζητά κανεί άλλο το λόγο σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Να σας υπενθυμίσω ότι τον Νοέμβριο προβλέπεται ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Όπως είπε η κυρία Μάισνερ, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα πρέπει να δούμε αν ε, στα πλαίσια του τριμερού διαλόγου θα μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να επανέλθουμε στον προπολογισμό για το 2012. Δεν έχει έρθει ο εισηγητής, αλλά να σας διαβάσω αν είδη εισαγωγή στις σημειώσεις του Πρόεδρου. Και άμα έρθει ο συγγετής, θα συνεχίσει αυτός. 54 τροπολογίες οι οποίες καταθέτηκαν. Δύο γραμμές του προπολογισμού και 17 του εισηγητή. Επιπρόσθετα, 13 τροπολογίες για το σχέδιο της ε, νομοδότησης Υπό τη νέα διαδικασία, η θέση του Κοινοβουλίου, η οποία θα υιοθετηθεί το Οκτώβριο, θα προσαρμοστεί σε αυτή του Συμβουλίου μέσω Επιτροπής Συνδιαλλαγής. Και αυτό θα επιτρέψει την έγκριση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Οι θέσεις του Συμβουλίου περιλαμβάνουν μείωση περίπου 1,6 δις ευρώ σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις τις υποχρεώσεις και 3,6 δις σε ό,τι αφορά τις πληρωμές συμπεριλαμβανομένης μείωσης 140 εκατομμυρίων και πλέον σε ό,τι αφορά τις πληρωμές για την πολιτική για τις μεταφορές. Αυτό συνοδεύεται και από μια διακήρυξη, μια δήλωση που καλεί από την Επιτροπή, στην Επιτροπή να καταθέσει ένα τροποποιημένο προπολογισμό σε περίπτωση που δεν επαρκούν αυτές οι περικοπές. Ο εισηγητής προτείνει πολλές από αυτές τις περικοπές να τις αναρέσουμε, επικεντρωνόμενος στις πολιτικές προτεραιότητες που έχει θέσει η Επιτροπή. Επίσης, ο εισηγητής προτείνει ε, τροπολογίες για να διασφαλιστεί ότι οι εξωτερικέ υπηρεσίες έχουν επαρκές προσωπικό για να εκτελέσουν τις νέε τους υποχρεώσεις. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω στην παρούσα φάση. Και θα δώσω το λόγο στους ομιλητές από τις ομάδες. Αν έρθει ο κ. Λιμπεράτσκι θα του δώσω το λόγο. Αλλά να αρχίσουμε καταρχάς από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είπατε και τα νούμερα και τα βασικά. Κατά άποψή μου, στην πραγματικότητα υπάρχει μια μεγάλη σύγκληση απόψεων μεταξύ του εισηγητού και των σκιώδων εισηγητών από τις διάφορες ομάδες. Ο προπολογισμό όπως ε, υποβάλλεται από το Συμβούλιο και όπως τροποποιήθηκε από την Επιτροπή έχει σχετίζεται με μια πολύ σημαντική πολιτική συζήτηση. Σε μια κρίσιμη περίοδο χρειαζόμαστε περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη. Χρειάζεται να προσαρμόσουμε τις φιλοδοξίες μας στα, μέ... στα μέσα μας ή να ανεβάσουμε τα μέσα μας στο επίπεδο των φιλοδοξιών μας. Εμείς ε, παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς μαζί με τον κύριο Λιμπεράτσκι που μπαίνει μέσα και θα τον ε, βοηθήσουμε σε όσες προσπάθειες καταβάλει για να βελτιώσουμε εκ νέου τον προπολογισμό στα αναγκαία, λαμβάνοντας υπόψη και εδώ πρέπει να τονίσουμε την υφιστάμενη πραγματικότητα. Δεν θα προτείνουμε ένα ε, εικονικό ή ονειροπαρμένο προπολογισμό, αλλά ένα ρεαλιστικό, σοβαρό προπολογισμό. Αυτό είναι κάτι που το θέλουμε όλοι στην Επιτροπή. Οι μεταφορές είναι βασικό κομμάτι των ευρωπαϊκών πολιτικών και της ικανότητας να ε, αντιμετωπίσουμε την κρίση με βέβαια υφιστάμενο το ζήτημα της σύγκρουσης ε, με τον διακυβερνητισμό και το ότι οι οργανισμοί θεωρούνται διακυβερνητικά όργανα ε, που αποτελούν, εγώ πιστεύω ωστόσο ότι αποτελούν ε, ένα βασικό εργαλείο της πολιτικής μεταφορών. Υπάρχει λοιπόν εν γέννη μεγάλη σύγκληση απόψεων και επί της ουσίας και επί των τοπολογιών με αυτά που είπε ο εισηγητής και βλέπουμε ότι πολλές τοπολογίες μάλιστα μπορούν να συγχωνευτούν και πιστεύω ότι θα υπάρχει αρκετά μεγάλη συμφωνία στην Επιτροπή μα στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ. Κύριε Λίτμπεράτς και εγώ εξήγησα πριν μπείτε τις 54 τροπολογίε που υποβλήθηκαν, τις 17 δικές σας, τις 13 για το σχέδιο γνωμοδότησης. Επίσης τόνισα προς την Επιτροπή ότι το Συμβούλιο προτείνει τεράστιες περικοπές στον προπολογισμό εσείς προτείνετε να επαναφέρετε τις περικοπές με έμφαση στις πολιτικές μας προτεραιότητες. Δεν ξέρω αν θέλετε να λάβετε το λόγο τώρα. Απάντησε ο κύριος Ρικέ. Νομίζω ότι ακούσατε τα περισσότερα από αυτά που είπε. Μετά θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους κύριους. Ο κύριος και έχει το λόγο τώρα όμως. Πρόεδρε, Συγγνώμη που καθυστέρησα καταρχά. Από ό,τι κατάλαβα, να τα πω στα αγγλικά. Έλεγα λοιπόν, συγγνώμη που καθυστέρησα. Είχαμε μια επιμήκυνση του χρόνου δουλειά στην ομάδα εργασία. Αυτό που άκουσα από τον κύριο Ρικέ αντικατοπτρίζει και το πνεύμα της ομάδας εργασίας και με τους σκιώδεις. Τρία ζητήματα, τρεις ομάδες ζητημάτων έχουμε. Πρώτον, μια μείωση 140 εκατομμυρίων ευρώ από πλευράς του Συμβουλίου. Εμείς διαφωνούμε με αυτό γιατί πρόκειται για δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικού χαρακτήρα αλλά που θέλουν να δώσουν κίνητρα και ανάπτυξη εθνικό επίπεδο, άρα και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Συμφωνήσαμε λοιπόν και με τους κύριους συζητητές ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι αρχι... τα αρχικά κονδύλια όπου υπέβαλε και η Επιτροπή. Δεύτερον, τα πιλωτικά σχέδια. Ως εισηγητές ετοιμάσαμε έξι πιλωτικά σχέδια. Καταγράψαμε τη θέση των συντονιστών στις 23 Μαΐου του 2011. Τρία από τα έργα αυτά θα συνεχιστούν για λόγους τεχνικούς ή διαδικαστικούς, ενώ κάποιες τροπολογίες αφορούν ακριβώς τα έργα αυτά. Πρέπει είναι οι τροπολογίες της κυρίας Τικάου με την οποία μίλησα, αλλά και της κυρίας Αγιάλα Σέντερ που συζητήσαμε επίση στις ομάδες εργασία. Η τρίτη ομάδα ζητημάτων που είναι σημαντική για μας είναι οι επιμέρους προτάσεις που θέλω τάχει να παρουσιάσω. Υπάρχει ένα λάθος καταρχάς. Η τροπολογία 6.727 πρέπει να είναι μία τροπολογία. Ζητώ λοιπόν να την διορθώσετε. Σε ό,τι αφορά το 6751, 67 και 52 και 53 για τους λόγους που προανέφερα και που συζητήσαμε ε, λόγω έλλειψης νομικής βάσης προτείνω να, την, να τις κατοψηφίσουμε. 6.713 τυραν τώρα, τυπικά, πρέπει να απορριφθεί, γιατί εδώ η κυρία Ντιράν προτείνει μια ποσόστοση 0-0, δηλαδή να περάσει ένα πολιτικό μήνυμα. Αυτό θέλει η κυρία Ντιράν, ώστε στους επόμενους προπολογισμού ο κλάδος αυτός να καλυφθεί. Με αυτή την αιτιολόγηση θα δεχόμουν την τροπολογία. 6707. Δαντάν και λοιπόν αφορά τον σιδηροδρομικό οργανισμό, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Εγώ προτείνω να απορριφθεί η τροπολογία αυτή, διότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων είχε μια χαμηλή αξιολόγηση κυρίως λόγω χαμηλών δαπανών. Υπάρχει επίσης και το rate of error, το επίπεδο σφάλματος. Κατά συνέπεια, θέλουμε τυπικά να ε, επαναφερθεί στην τάξη. Κατόπιν, τροπολογία άλλα Σέντερ και Νταμέντι αφορούν και αυτές τα πιλωτικά προγράμματα. νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσουμε να τα δεχθούμε, αλλά αυτό είναι εξαρτάται από εμά. 67-14. το τροπολογία που προτείνει τουρισμό με σιδηρόδρομο, δηλαδή μια σιδηροδρομική δραστηριότητα τουριστικού χαρακτήρα που μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα ε, πρόταση σε μια περίοδο κρίσης, προτείνω ωστόσο να απορριφθεί ε, το, για τις τροπολογίες τη γνωμοδότηση. Η έξι της κυρίας Τυρνό ε, θα πρέπει να τη διευκρινίσει κύριε Τυρνό. Δεν καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται και κατά συνέπεια δεν μπορώ να πω αν είμαι υπέρ ή κατά. Τροπολογία 9 τώρα. του κύριου Μπαλτσίτης. Θεωρητικά είναι σωστή η τροπολογία, αλλά δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, δική μας ευθύνη. Άρα προτείνουν την απόρριψη. Τροπολογία 11 είναι απορριπταία, ενώ η 13 και Βλαστό γροστατα προτείνει την διαγραφή της λέξης σόφρον, φρόνιμη χρηματοδότηση. Εγώ την δέχομαι, χωρίς ωστόσο τον όρο prudent, σόφρον, που αποδυναμώνει το υψηλό επίπεδο στάνταρτ που έχουμε θεσπίσει. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους και όσους έχουν υποβάλει απολογίες περιμένω τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρικέ να προσθέσει κάτι. Δύο λόγια για το 6707 των Σιδηροδρομικό Οργανισμό. Να επαναλάβω προς τον συνάδελφο Λιμπεράτσικη ότι ο Ευρωπαϊκό Ιδεοδομικό Οργανισμός είναι σε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση και την ξέρω γιατί είμαι κοντά στην υπηρεσία. Έχει μια αύξηση, συνεχή αύξηση των ευθυνών που τις ανατίθενται χωρίς αύξηση των πόρων που τις διατίθενται. Η δημιουργία ενός οργανισμού όπως αυτού που μπορεί να εξελιχθεί δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων. Καταλαβαίνω η παρατήρηση του κ. Λιμπεράτσκι είναι σωστή. Όντως έχουν γίνει παρατηρήσει που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν θα ήθελα πολιτικά ωστόσο να αποδυναμώσουμε τον οργανισμό, αλλά να τον βοηθήσουμε να ενισχύσει το ρόλο του. Ξε, ξέρουμε ότι ο στόχος πάντων, των αντιπάλων του διακυβερνητισμού είναι η αποσταθεροποίηση των εξωτερικών υπηρεσιών και οργανισμών. Αλλά καταλαβαίνω τα σχόλιά σας, αλλά πολιτικά θα, δεν θα ήταν σκόπιμο να, την, ε, να αποδυναμώσουμε τον οργανισμό αυτό ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, συμφωνώ με τις παρατηρήσεις, αλλά ήθελα να δείξουμε ότι σκεφτόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτός ο οργανισμός. Ευχαριστώ. Κύριε Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Λιμπεράτσκι που επεξεργάστηκε αυτό τον προϋπολογισμό. Είπε ότι σε πολλά πράγματα συμφωνούμε, χρειαζόμαστε για τις μεταφορές λεφτά οπωσδήποτε, αλλά πρέπει να είμαστε λογικοί στα αιτήματα και στις δαπάνες και εμεί είχαμε νότητα γιατί όταν ήθελε να περικόψει η Κομισιόν όλοι μαζί θελήσαμε να αποκαταστήσουμε την κατάσταση ε, και για τους οργανισμούς αποκτήσαμε αυξημένες ευθύνες ε, αν σκεφτείτε τους ενιαίους ουρανούς ή το πρόβλημα ε, ρήπανσης ε, ε, οι αρμοδιότητες των οργανισμών εδώ αυξάνονται και δεν μπορούμε να περικόπτουμε και για τα πιλωτικά συμφωνήσαμε, το είπε ο εισηγητής, θέλουμε ενιαία να τα συστήσουμε και να τα διατηρήσουμε και για την βιομηχανική κληρονομιά, κοιτάω τον πρόεδρο εδώ, τον τουρισμό με πρόσβαση για όλους και την ε, ενιαία κράτηση ε, στις μεταφορές. Αυτό μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Η ομάδα μας η ίδια έκανε παρατηρήσεις μόνο σε θέματα που εγκρίνονται με μεγάλη ομοφωνία. Δεν θέλουμε να αυξηθούν πολλοί οι ε, Θα επισέλθω σε ορισμένα πράγματα όμως για να πω τη στάση που θα κρατήσουμε. Για την κυρία Τικάου για τους ευρωπαϊκούς προορισμούς αριστείας. Αυτό θα πρέπει να υπάρχει στον τουρισμό, να αναπτυχθεί δύο εκατομμύρια θέσεις, αλλά εδώ δεν θα συμφωνήσουμε παρόλο που είμαστε υπέρ του τουρισμού. Ε, είναι υπερβολικό ήδη, θέλουμε να κάνουμε πολλά για τον τουρισμό, αλλά θα πρέπει να είναι σόφρον η ε, δημοσιονομική μας προσέγγιση. Εδώ θα ψηφίσω λοιπόν. Θέλω επίσης να πω, είπα προηγουμένως λίγα πράγματα, είναι πολύ ωραίο να πούμε ότι χρειάζεται ε, σχολή για να μαθαίνουν τα παιδιά το ποδήλατο και να είναι ασφαλής. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα αυτή την εποχή. Δεν επαρκούν για όλη την υποδομή και τη βελτίωσή της στην Ευρώπη. Εγωιτευτική ιδέα, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αυτά είναι τα βασικά που ήθελα να αναφέρω. Σταματώ εδώ προς το παρόν. Γενικά νομίζω ότι είναι πολύ σόφρονο πυροπολογισμό και πολλά αύριο επίσης θα μπορέσουν να ψηφιστούν ομόφωνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζέλλερ. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Λιμπεράτσκι για όλη αυτή τη δουλειά που έκανε. Ως εκπρόσωπος του ομάδας ECR στην Επιτροπή Μεταφορών δεν μπορούμε 100% ε, να προσυπογράψουμε το σχέδιο έκθεσης. Εξακολουθούμε βέβαια να εκτιμούμε όλος ιδιαίτερος το έργο σας. Ε, από πολιτική πλευρά καταλαβαίνουμε το κίνητρο γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εις ό,τι αφορά τις πιστώσεις ε, και τις πληρωμές που αναφέρεται στη θέση του Συμβουλίου. Σε πολλές χώρες η δημοσιονομική κατάσταση είναι αρκετά σφιχτή. Ιδιαίτερα αυτό έχει να κάνει τους οργανισμούς όπου πρέπει να επανέλθουμε στο σχέδιο του πρόταση του Συμβουλίου και να αυξήσουμε την ικανότητά τους. Ορισμένα μέλη εξακολουθούν να πιστεύουν και να στηρίζουν αυτές τις γραμμές, δηλαδή την αύξηση Τέντη, Μάρκο Πόλο 2 και τη γραμμή εκείνη που αφορά την πρόταση της Κομισιόν για πληρωμές και υποχρεώσεις ε, και ε, στο πρόγραμμα ΣΥΖΑΡ. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση, παρόλο που μπορούμε να συζητήσουμε ακόμη για αυτές τις γραμμές του προϋπολογισμού. Το ίδιο ισχύει και για τα περισσότερα πιλωτικά έργα. Απ' τη μια γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητα, ε, χρήσιμα τα πιλωτικά έργα, αλλά από την άλλη πλευρά πολλές φορές τα πιλωτικά έργα δεν εκπληρούν τους στόχους που έχουν τεθεί. Το λέω και εκ Θα εξηγήσω και πάλι την ε, θέση της ομάδας μου. Η πολιτική ομάδα από πίσω, η πολιτική ιδέα είναι ότι είναι δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ, κυρία Ντουράν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την εργασία του. Θέλω να διευκρινίσω κάτι, γιατί υπάρχει μια ερώτηση σε μια τροπολογία. Την τροπολογία 6 πρέπει να καταλάβουμε τι εννοείται. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προάγουμε τις επενδύσεις για την καταπολέμηση του θορύβου, αλλά και το RTMS και το τροχαίο υλικό και την υποδομή πρέπει να δούμε, γιατί συχνά επενδύουμε στον ένα και όχι στον άλλο τομέα και μετά δεν έχουμε ε, διασφαλίσεις ε, ασφάλειας. Ε, και τα δύο πρέπει να τα δούμε μαζί. Περί αυτού πρόκειται. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή που μίλησε και υποστήριξε την έννοια του αηφόρου βιώσιμου τουρισμού. Θα μιλήσουμε για αυτά όταν μιλήσουμε για τουριστικά στατιστικά στοιχεία για να προωθήσουμε όλους τους τομείς που θα κάνουν να ανθίσει ο τουρισμός, να μειώσουν το διευσίδιο του άνθρακα, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας κλπ. Στην τροπολογία 4 δεν θα εκπλαγείτε ε, που σας ζητάμε να στηρίξετε μια τροπολογία που θέλει να διοχετεύσουμε κονδύλια στις ε, ε, υποδομές των μεταφορών. Αυτό είναι κάτι που λαμβάνει υπόψη το εξωτερικό κόστος. Όταν επιλέγουμε τις επενδύσεις πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα επιλέξουμε επενδύσεις που θα οδηγούν σε περιορισμένο εξωτερικό κόστος. Δεν θέλουμε δηλαδή να ε, αυξηθεί περισσότερο το κόστος ε, στην πορεία. Και μετά είναι και η τροπολογία η τρίτη, υπαριθμών 12 μετά το, για μετά το 2012 που πρέπει να φροντίσουμε ότι δεν θα αφαιρεθούν πόροι από τον τουρισμό. Αυτό έχει να κάνει με τις ε, δράσεις που είχε υπόψη να κάνει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Κυρία Γιάλα Ζέντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λιμπεράτσικε για το ενδιαφέρον που έδειξε στην εξέταση και ανάλυση των τροπολογιών ακόμα και εκείνων που δεν αποτέλεσαν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι και απλά μέλη του Κοινοβουλίου να είμαστε μπορούμε να συνεχίσουμε να υποβάλουμε τροπολογίες με κάποια βιώσιμη ελπίδα να τύχει της υποστήριξης των συναδέλφων παρότι δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των σκιωδών εκ των προτέρων να μιλήσω για δύο τροπολογίες. Πρώτον, πιλωτικά σχέδια, δεύτερον, προπαρασκευαστικά έργα, προπαρασκευαστικές πράξεις. Για το πρώτο, αυτό που λέω δεν είναι να φτιάξουμε ένα σχολείο υπόδομη, απλά η νέα λευκή βίβλος δίνει την ε, όθηση για μια ευρωπαϊκή πολιτική στην, στις αστικές μεταφορές ιδίω τη χρήση ποδηλάτου. Στην Ισπανία που υπάρχει πραγματικά boom κυκλοφορία ποδηλάτων υπάρχουν ορισμένε, ε, συγκρούσει μεταξύ πεζών και ποδηλατών. Θέλουμε λοιπόν μέσω προγραμμάτων που ενδιαφέρουν τα σχολεία να περάσουμε την ποδηλατική κουλτούρα Γι' αυτό είπα και εγώ, γι' αυτό το πολύ περιορισμένο μικρό πιλωτικό σχέδιο που δεν έχει μεγάλη επίδραση στον προπολογισμό και που πήρε το πράσινο φως από την Κομισιόν. Θα ζητούσα λοιπόν, θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να το λάβουν υπόψη. Δεν είναι εύκολο να δεχθεί πιλωτικά σχέδια του Κοινοβουλίου η Κομισιόν. Το έκανε σε αυτή την περίπτωση. Άρα καλό θα ήταν να μπορούσε η Επιτροπή να δεχθεί την πρότασή μας. Μετά, το δίκτυο δικής ασφάλειας. Παλιό έργο, παλιό σχέδιο που δεν έχει υποστηρίξει μέχρι τώρα η Επιτροπή. Τώρα το υποστηρίζει. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά φαντάζομαι ότι οι διαπραγματεύσεις που είχαμε για την οδηγία για τις κλήσεις, ε, για τα πρόστιμα, ε, ενίσχυσε την δημιουργία δικτύων μεταξύ ενώσεων θυμάτων, ε, βοηθά την Επιτροπή νομίζω και το Κοινοβούλιο, ώστε να κάνει ένα λόμπι για την ασφάλεια, την οδική ασφάλεια. Κοιτάξτε, δυσκολεύομαι πολύ να μιλάω όταν μιλάτε κι εσείς, έτσι. Πάντως, Αντί για συγγνώμη Ματέος, να υποστηρίξει το υπολογισμό, οπότε θα είμαι πανευτυχής για αυτή την κουβέντα που κάνετε μεταξύ Βελγίου Ιταλίας. Θα ζητούσα από, τους, από τις ομάδες, την κυρία Μάισνερ, να υποστηρίξουν τους υπολογισμού. Λεφτά πολλά δεν έχει. Η Κομισιόν είναι υπέρ, είναι θετικές πρωτοβουλίες, γιατί δεν τις ψηφίζετε. Κύριος Μπραντμπορν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφο ήταν πολύ διπλωματικό στην απάντησή του. Δεν θα είμαι εξίσου διπλωματικό, εγώ πολύ φοβάμαι. Θα ήθελα να κάνω κάποια γενικά σχόλια και μετά να περάσω σε κάποιε πιο ειδικέ παρατηρήσει για το κείμενο που έχουμε μπροστά μα. Καταρχά, θα ήθελα να πω ότι κάθε χρόνο δεν καταλαβαίνω πού βρισκόμαστε. Γιατί έχουμε προτάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίε είναι μη Και μετά ακόμα πιο πολύ μη ρεαλισμός μαζεύεται από την Επιτροπή μας σε ό,τι αφορά τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Σε ποιο πλανήτη ζούμε, ρωτιέμαι. Όλα τα κράτη-μέλη αναγκάζονται να κάνουν περικοπές στον προπολογισμό τους. Όχι επειδή το θέλουν, επειδή αναγκάζονται. Το ίδιο ισχύει στην Ισπανία, στον Εμένο Βασίλειο, στην Ιταλία, παντού. Και εμείς εδώ ζητάμε όχι μόνο να αναιρεθούν οι περικοπές που έχουν γίνει, αλλά να αυξηθεί ο προπολογισμό της ε, Επιτροπής μας. Νομίζω ότι ζούμε στο δικό μας πλανήτη, Πρόεδρε, και θα πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Δεν μιλάμε για τα ευρωπαϊκά χρήματα, μιλάμε για χρήματα του φορολογούμενου και ο φορολογούμενος αναγκάζεται να καταβάλει όλο και πιο πολλά εν είδη φορολογίας για να καλύψει τα ελλείμματα στα κράτη-μέλη, τα εκάστοτε. Γιατί θεωρείτε ότι θέλει ο φορολογούμενος να δώσει πιο πολλά χρήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάποια συγκεκριμένα σχόλια τώρα για την θέση στην οποία βρισκόμαστε και Προφανώ, από καταλαβαίνετε, υποστηρίζω την θέση του Συμβουλίου και αυτή θα ήθελα να επικρατήσει. Αλλά σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες, ε, τα συγκεκριμένα στοιχεία, χαίρομαι που ο κύριο Λιμπεράτσκι αναγνωρίζει ότι, για παράδειγμα, στην τροπολογία 9 στην γνωμοδότηση πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, αυτή τη δική μας επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διαγράψουμε αυτή την τροπολογία, γιατί θεωρώ ότι είναι και κακή ιδέα, άλλωστε. Δεύτερο στοιχείο. Νομίζω. Για την τροπολογία 13. Δεν ναι, πίστευα στα μάτια μου όταν είπα την τροπολογία αυτή. Θέλουμε να βγάλουμε τη λέξη σόφρον σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των οργανισμών. Τι θέλουμε, τη δηλαδή, λένε μη σόφρον. Η χρηματοδότηση. Να ξοδεύουν τι θέλουν. Αυτό είναι παλαβό θεωρώ. Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, Πρόεδρε, επιτάσσει σοφροσύνη και χρειαζόμαστε ε, περικοπές όπου δεν είναι απαραίτητες, ε, απαραίτητη χρηματοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε σε ό,τι αφορά την προσέγγιση μας, γιατί δεν εξετάζουμε project τα οποία δεν ε, αποτελούν πλέον προτεραιότητα ή επίσης δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας. Γιατί δεν μεταφέρουμε λοιπόν χρήματα από τέτοια project σε project που είναι πιο ελπιδοφόρα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειαστούν να αυξηθεί ο προπολογισμό. Θα γίνονταν περικοπέ, μάλιστα. Και αυτό φαίνεται ότι δεν το πήραμε υπόψη σε καμία διαπραγμάτευση ως τώρα. Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι τελείως μη ρεαλιστική αυτή η προσέγγιση μας. Ποτέ δεν θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε ούτε με την Επιτροπή Προϋπολογισμού, ούτε με το Συμβούλιο σε επίπεδο συνδιαλλαγής. Δεν πρόκειται να μας δώσουν πιο πολλά χρήματα και αυτό είναι σαφές για όλα τα κρατημέλη. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομη παρατήρηση προς τον συνάδελφο Μπράντμπερν. Αφήνω γενικότερο, γενικότερα το βρετανικό θέμα, αλλά όταν τα κράτη-μέλη όλο και περισσότερο ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες και θέλουν αυτό να γίνει με περικεκομένο προϋπολογισμό, ε, τότε θα είναι μεγάλη η πολεμική που θα αναπτυχθεί και που κανείς δεν τη θέλει. Οι οργανισμοί έχουν ένα σημαντικό καθήκον να παρακολουθούν, να εποπτεύουν, να μετεξελίσσουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες ώστε να είναι οι σωστοί. Και θα πρέπει να τους τη δώσουμε την ευκαιρία να το κάνουν αυτό. Γιατί αν περιοριστούμε ε, στα κοντήλια αυτό δεν θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της Ένωσης. Κάτι άλλο ακόμα να συμπληρώσω και να διευκρινίσω τον, την προαγωγή του σιδηροδρομικού τουρισμού και τη πεζοπορία, τη χρήση ποδηλάτων κλπ έχω υπόψη μου κάτι που προέρχεται πολύ και από τους ίδιους τους επιβάτες που λένε ένα μεγάλο έλλειμμα είναι ε, η διοικητική διεκπαιρέωση των αποσκευών. Όλη αυτή η αλυσίδα των αποσκευών και του χειρισμού. Είναι μεγάλα τα εμπόδια εδώ για το σιδηροδρομικό τουρισμό, τις μεταφορές τουριστών με σιδηρόδρομο σε σχέση με άλλες. Μπορούμε λοιπόν εδώ να διευκρινίσουμε κάτι, να προσθέσουμε δηλαδή ε, βελτίωση της πολυτροπικής διεκπαιρέωσης των αποσκευών, κάτι τέτοιο, για να αντιδράσουμε σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο το θέτουν οι επιβάτες και οι οργανώσεις τους. Και πολλοί μας ρωτούν ε, γιατί δεν ε, ε, προάγεται το θέμα αυτό. Γι' αυτό άλλωστε προτιμούν να πάνε με γιοταχή... Ε, στα ταξίδια τους από ό,τι με το σιδηρόδρομο. Είναι ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, αν θελήσουμε δηλαδή να μπούμε στις λεπτομέρειες. Ο κύριος Κόσμαν από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστήσουμε την Επιτροπή και τον εισηγητή για τη γενικότερη υποστήριξη στις προτάσεις της Κομισιόν και όπως είπατε οι περισσότερες τροπολογίες που προτείνουν θέλουν να αποκαταστήσουν τις πιστώσεις ε, στο ύψος του προϋπολογισμού του 2012 και αυτό το χαιρετίζουμε γιατί διατηρούμε την εφαρμογή της ε, πολιτικής μας και να διατηρήσουμε την ε, εκτέλεση των έργων. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν την Επιτροπή για το έργο της και προσβλέπω με ενδιαφέρον στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λιμπεράτσκι έχει να προσθέσει τίποτε. Ευχαριστώ. Ε, εμείς ε, είμαστε πεπισμένοι, κύριε Μπράντμπορν, ότι δεν έχουμε εδώ ε, παράλογα έργα αυτός ε, ο τρόπος εκτέλεσης ή και ε, κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι διαφορετικός. Δεν θέλουμε ε, να κάνουμε περικοπές πάση και πάμε στο αρχικό μας μήνυμα. Θέλουμε να δημιουργηθούν καινούριε δυνατότητες και ευκαιρίε μέσα από την έγκριση του προπολογισμού. Και προκειμένου περί των κάποιων συγκεκριμένων ε, θεμάτων που σχολιάστηκαν, ιδιαίτερα την ε, τροπολογία 6, ε, άκουσα πολύ προσεκτικά την, ε, την εξήγηση της κυρίας Ντουραν, αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά την υποδομή να την φροντίσουμε και όχι να μιλάμε για τις αγορές τροχαίου υλικού κλπ. Δεν είναι αυτή η ώρα. Ε, δεν θα πρέπει δηλαδή να ε, ασχοληθούμε εμείς με αυτό. Όταν πρόκειται τώρα για τον οργανισμό, τον, ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, έχουμε εδώ ένα εκατομμύριο δεσμευμένο Συνολικά ε, έχουμε δηλαδή εδώ το 6% του προϋπολογισμού, περίπου 16 συνολικά είναι τα εκατομμύρια. Πάμε στις επιφυλάξεις. Ε, φτάσαμε πολύ κοντά να μην χορηγήσουμε απαλλαγή στον οργανισμό σιδηροδρόμων λόγω του μεγάλου χάους που επικρατούσε στον προϋπολογισμό αν γνωρίζετε καλύτερα το έργο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων και αν μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι αυτό είναι μόνο ο ελίπων κρίκος και κάποια κονδύλια που θα συμβάλλουν ε, στην καλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, εναδεχτώ το επιχείρημά σας. Και στρέφομαι τώρα στους συναδέλφους ε, ε, της πολιτικής μου ομάδας για να ψηφίσουν υπέρ. τώρα, οι καιροί είναι δύσκολοι, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα ε, λογικά, τα ορθολογικά ε, έργα στη πολιτική των μεταφορών και επίσης θέλω να πω ότι οι μεταφορές δεν είναι... Ε, δεν ενδείκνυται ως τομέας για να κάνουμε περικοπές είναι ένας τομέας ο οποίος δίνει έναυσμα για περαιτέρω ανάπτυξη και δραστηριότητες στις επιχειρήσεις. Ελπίζω να συμφωνούμε σε αυτό και να συμφωνήσουμε ε, να επανέλθουμε στα ποσά που αρχικά είχε προτείνει η Κομισιόν και που δεν ήταν και πολύ υπερβολικά. Πάλι ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ευγενικά για την προσοχή σας και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους ε, για την ε, θετική του στάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λιμπεράσκη. Να σας πω το χρονοδιάγραμμα. Ψηφίζουμε αύριο στην Επιτροπή. Κατόπιν η Επιτροπή Προεπλογισμών θα ψηφίσει 4 με 6 Οκτωβρίου. Θα περάσει στην Ολομέλεια όλος ο προϋπολογισμός, στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Αύριο ψηφίζουμε, Ολομέλεια Οκτώβριος. Ευχαριστώ. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ανταλλαγή απόψεων για τον πίνακα αποτελεσμάτων για την καταναλωτική αγορά. Ανταλλαγή επιτροπών με την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ τη επιτροπή. Η κυρία Τίλεν είναι εδώ, αναπληρώτρια επικεφαλής ε, διευθύντρια που θα σχολιάσει τις ε, αρχικές συζητήσεις, θα κάνει την εισαγωγή μάλλον. Ο συνάδελφος προσπαθεί να στήσει την παρουσίαση για να παρακολουθείτε ευκολότερα αυτά που θα σας πούμε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας επιτρέψετε να παρουσιάσουμε τις εργασίες για την παρακολούθηση αγοράς και των πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη δουλειά αυτή στην Επιτροπή. Θα ξεκινήσω δίνοντάς σας το πλαίσιο της δουλειάς αυτής. Στην Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ τέσσερα χρόνια σχεδόν πριν ξεκινήσαμε να συλλέγουμε δεδομένα που εξετάζουν τη λειτουργία των αγορών από την οπτική γωνία του καταναλωτή. Επίσης αναλύσαμε τις δυσλειτουργίες ε, της αγοράς και τις προτινόμενες αλλαγές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε την αγορά από την ε, οπτική του καταναλωτή, ούτως ώστε να μην βλέπουμε μόνο ζητήματα της προσφοράς και θέματα ανταγωνισμού, αλλά να τα δούμε και από τη μεριά του καταναλωτή. Ιδίω δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να επιτρέψουν καλύτερη λειτουργία της αγορά, Διότι πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές έχουν ε, και τα εργαλεία και τι δυνατότητε να καταλάβουν αυτούς τους, ε, τις σύνθετες επιλογές που αντιμετωπίζουν. Μιλάμε για καινοτόμες υπηρεσίες που βοηθούν τον ανταγωνισμό. Πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο αυτό και για τους πολιτικούς ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Τα στοιχεία μπορούν να συστοιχίσουν την επίδοσή τους σε σχέση με άλλων κρατών μελών, επιτρέποντας ε, να αλλάξουν τα, τα προβλήματα, τα βασικότερα προβλήματα σε κάθε χώρα. Να σας πω τι στοιχεία συλλέγουμε και τι εργαλεία αναπτύξαμε. Ο στόχος μας είναι ο πίνακα αποτελεσμάτων για του καταναλωτέ, που είναι ένα σύστημα προειδοποίηση που πληροφορεί του ε, πολιτικού ε, για τα προβλήματα τη αγορά. Κάθε χρόνο έχουμε δύο, δύο, εκδίδουμε δύο τέτοιους πίνακες, έξι μέχρι τώρα έχουμε και έχουμε δύο κατηγορίες ε, πίνακα. Την άνοιξη είναι οι συνθήκες καταναλωτή όπως τις λέμε, που είναι ένας πίνακας που εξετάζει δύο τομείς. Την ενσωμάτωση του ιανεμπορίου στην εσωτερική αγορά, δηλαδή βλέπει διασυνοριακά ζητήματα και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και δεύτερον, το ανοιξιάτικο, ο ανοιξιάτικος πίνακας, εξετάζει το εθνικό, τις συνθήκες και το περιβάλλον στα κράτη-μέλη, σε κάθε κράτος μέλος. Το φθινοπορεινό, που το λέμε αγορά κατανο... πίνακας αποτελεσμάτων αγοράς ε, καταναλωτή, βλέπει τις, πιθανό... τις πιθανές δυσλειτουργίες των αγορών, παίρνουμε κάποιες αγορές και τις βάζουμε σε σειρά ανάλογα με το πόσο καλά λειτουργούν για τον καταναλωτή πάμε και ένα βήμα παραπέρα στην ανάλυση αυτή. Επιλέγουμε μία ή δύο αγορές από τις κακές για να μπούμε λεπτομερέστερα στην ανάλυση τους και να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής στις αγορές αυτές. Πίνακας των καταναλωτικών, ε, των αγορών για τον καταναλωτή όπως σας είπα βγαίνουν το φθινόπωρο. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε είναι ένα, μια ετήσια έρευνα της αγοράς 50 καταναλωτικών αγορών. Ζητούμε την άποψη του καταναλωτή για αυτές τις 50 αγορές, για τα 50 είδη. Επιπλέον εξετάζουμε το θέμα της τιμολόγησης, την μεταβολή των τιμών κυρίως μεταξύ κρατών μελών και τις καταγγελίες από πλευράς καταναλωτών. Η έρευνα αυτή, παρακολούθηση της αγοράς, που είναι η βάση του πίνακα αποτελεσμάτων, εξετάζει τις αγορές. Πρώτη φορά την κάναμε την έρευνα αυτή πέρσι και τα αποτελέσματα είναι στο τέταρτο, στη τέταρτη έκθεση. Έφερα και κάποια αντίγραφα από αυτά τα scoreboards, αν τα θέλετε, που βρίσκονται στην είσοδο του Τη αίθουσα ε, στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσε, αν τα αγγλικά δεν είναι εύκολη γλώσσα για εσά. 50 αγορέ, λοιπόν, 50 προϊόντα που είναι περίπου 60% των δαπανών του καταναλωτή. Η έρευνα τον πρώτο χρόνο έγινε και στα 27 κράτη-μέλη σύν την Ορβηγία με συνεντεύξει με καταναλωτές που είχαν μόνο, μόνο με καταναλωτές που είχαν πρόσφατη εμπειρία με την αγορά. Γιατί θέλαμε την εμπειρία του, όχι την άποψή του την έρευνα τώρα την κάνουμε σε αιτήσια βάση για να, δούμε, για να βλέπουμε τάσεις. Αγορές, υπάρχουν κάποιες αγορές που πάνε καλύτερα και αυτό οφείλεται σε μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο. Οι, τα ερωτήματα που είχαμε στην πρώτη αγορά φορούν συγκρισιμότητα, εμπιστοσύνη, γενική ικανοποίηση, προβλήματα, καταγγελίες και ποιες αγορές χρειάζονται αλλαγή, switching. Ζητούμε από τους καταναλωτές να βαθμολογήσουν από το 0 έως το 10 μία αγορά. Φερρυπίν, στη συγκρισιμότητα λέγαμε από το 0 προς 10 πείτε μας πόσο δύσκολο ήταν να συγκρίνετε το προϊόν ή την υπηρεσία στην αγορά αυτή που πολλούσε είτε ο προμηθευτής είτε ο λιανέμπορος. Το ίδιο φορούσε, το ίδιο και για την εμπιστοσύνη. Από 0 προς 10 πόσο εμπιστεύεστε ότι οι έμποροι θα σέβονται τους κανόνες, θα σέβονται τους καταναλωτές, το ίδιο και η γενική ικανοποίηση. Ζητήσαμε επίσης από τους καταναλωτές να μας πούν αν το πρόβλημα, είτε με το, πρόβλημα, με το προϊόν ή την υπηρεσία, είτε με τον προμηθευτή ή τον λιανμπορό ε, που, πούλησε το προϊόν ή την υπηρεσία. Υπήρξαν καταγγελίες, ρωτήσαμε και όπως σας είπα, Ρωτήσαμε ιδιαίτερα ε, στις υπηρεσίες κοινή ωφέλεια αν άλλαξαν προμηθευτή, πόσο εύκολο ήταν. Επόμενο slide. Βγάλαμε τώρα ένα δίκτυ επίδοσης αγοράς για κάθε αγορά με βάση τα στοιχεία αυτά. Ο δείκτη περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία. Συγκρισιμότητα, εμπιστοσύνη, προβλήματα και καταγγελίε που τα εξετάζουμε από κοινού και γενική ικανοποίηση. Επίση, υπάρχει και ένα δεύτερο δείκτη, MPIS, Market Performance Indicator Switching, που έχει σημασία για τις αγορές όπου μπορεί να αλλάξει ο καταναλωτής προμηθευτή. Επόμενη διαφάνεια. Αυτή είναι η βαθμολογία, η σειρά που βγάλαμε, δεν ξέρω αν τη βλέπετε. 50 καταναλωτικών αγορών, όπως τις βγάλαμε μετά το MPI. Η σειρά που βλέπετε είναι η ευρωπαϊκή βαθμολόγηση, αλλά στο εθνικό, στο scoreboard έχουμε την ίδια βαθμολόγηση για κάθε μία εθνική αγορά. Οπότε μπορεί να δείτε πόσο καλά πάει η συγκεκριμένη αγορά στη δική σας χώρα. Σε αυτή την ευρωπαϊκή βαθμολόγηση δείτε ότι οι τρεις πρώτες καλύτερες αγορές για τον καταναλωτή είναι τα βιβλία, τα περιοδικά και εφημερίδες, οι προσωπικές ε, υπηρεσίες και η ψυχαγωγία και κουλτούρα. Οι τρεις χειρότερες αγορές είναι παροχή ίντερνετ, αγορά και επενδυτικές αγορές. Τώρα, αυτές που έχουμε στον κύκλο είναι αυτές που νομίζουμε ότι σας ενδιαφέρουν εσάς σαν Επιτροπή. Διακοπές, ξενοδοχειακή και στέγη, πάει καλά. Σιδηρόδρομοι και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, χαμηλά. Προτελευταίοι σχεδόν. Αλλά και η συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων είναι από τις πιο χαμηλές ε, σε ικανοποίηση αγορές. Στο μέσον βλέπουμε τις αεροπορικές εταιρείες, ταχυδρομικές υπηρεσίες courier, ενοικίες αυτοκινήτων, νέα αυτοκινήτα, αυτοκίνητα, ε, οργανωμένα ταξίδια, καύσιμα. Όπως σας είπα, αυτή η βαθμολόγηση των 50 αγορών υπάρχει και για κάθε κράτος μέλος. Το ίδιο γράφημα. Οπότε μπορείτε να δείτε και πώς είναι, ποια είναι η σειρά σε εθνικό επίπεδο κάθε αγορά σε σχέση με την ευρωπαϊκή, που είναι πολύ χρήσιμο για σκοπούς σύγκρισης και που το συζητούμε τακτικά με τις εθνικές καταναλωτικές αρχές και τις εθνικές αρχές επιβολής της νομοθεσίας, γιατί δείχνει που, ποιους τομείς πρέπει να προσέξει μια χώρα. Επόμενη διαφάνεια. Επίσης, έχουμε για κάθε αγορά τη σειρά αναχώρα. Εδώ βλέπετε πώς πήγε η βαθμολογία για τα οργανωμένα ταξίδια. Η Φιλανδία είναι καλύτερη, όπως βλέπετε. Τρεις χώρες έχουν πολύ χαμηλή βαθμολόγηση. Το σημαντικό είναι το εξή. Η απόκληση με μεταξύ της καλύτερης και της χειρότερης χώρας για τα οργανωμένα ταξίδια είναι 11 πόντι. Χαμηλότερο δηλαδή από το μέσο όρο άλλων αγορών. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τα οργανωμένα ταξίδια λειτουργούν με ομοιογενή τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, έχουμε και επιπρόσθετες πληροφορίες, όχι στο γράφημα αυτό, αλλά στο scoreboard για το πόσο καλά πήγαν οι αγορές σε σχέση με κάθε συνιστόσα του δίκτυ. Για την αγορά αυτή, τα οργανωμένα ταξίδια δηλαδή, βλέπουμε ότι η συγκρισιμότητα και η γενικότερη ικανοποίηση είναι κάπως ψηλότερα από το μέσο όρο, η εμπιστοσύνη είναι παρόμοια με το μέσο όρο, αλλά ο αριθμός των καταναλωτών που ανέφεραν ότι μετώπισαν προβλήματα είναι κάπως ψηλότερος από το μέσο όρο. Επόμενη διαφάνεια. Όχι. Να σας δείξω την ίδια διαφάνεια για μια άλλη αγορά που δεν πάει τόσο καλά. Σύμφωνα με την έρευνά μας. Τις συνδρομικές υπηρεσίες. Βλέπετε ότι η Λιθουανία και η Εστονία είναι καλύτερες, αλλά οι μισές χώρες περίπου δίνουν πολύ χαμηλή βαθμολόγηση το κενό, η απόκληση μάλλον στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταξύ του καλύτερου και του χειρότερου είναι 27,3 πόντι. Πάνω από δι, περίπου διπλάσιος ε, από το μέσο όρο. Άρα δείχνει μεγάλη απόκληση στην ε, επίδοση της αγοράς αυτής από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη. Αν δούμε προσεκτικότερα τις διάφορες συνιστώσεις αυτή της αγορά δηλαδή θα δούμε ότι παντού σχεδόν η αγορά πάει χειρότερα από το μισό Είναι δε εξαιρετικά χαμηλότερη και στη γενική ικανοποίηση και στα προβλήματα να βγάζει 2,5 φορές το μεσόωρο. Το ενδιαφέρον είναι ότι παρότι εμφανίζονται πολλά προβλήματα με την αγορά αυτή ε, από του καταναλωτέ, δεν παραπονιούνται συχνά. Next slide, please. Well, one, one last slide I, uh, or one last market I want to... Τελευταία αγορά που θέλω να σας δείξω. Αεροπορικές εταιρείες. Μια από τις ε, αγορές με τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των υπηρεσιών δικτύων που είναι αυτή η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του καταναλωτή και έχει καλύτερο σκορ και στη συγκρισιμότητα και στην εμπιστοσύνη. Εκεί όμως έχει προβλήματα, προβλήματα, προβλήματα πάνε χειρότερα από το μέσο όρο. Η απόκληση δε μεταξύ του καλύτερου και του χειρότερου είναι πολύ μικρή. Αυτό τι δείχνει. Πρόκειται για μια ομοιογενή, αρκετά ομοιογενή αγορά σε ό,τι αφορά την επίδοσή τη ανά την Ευρώπη. Επόμενη διαφάνεια. Αυτό σας δείχνει την εικόνα, μια πολύ μικρή εικόνα του πώς του πλούσιου περιεχομένου που έχει αυτό ο πίνακα αποτελεσμάτων. Προφανώ μπορούμε να σα δώσουμε όλα τα στοιχεία τώρα, αλλά έχουμε μια συνοδευτική έκθεση πολύ μεγάλη, με λεπτομέρειε, με ανάλυση για όλου όσου ενδιαφέρονται, ενώ περιγράφουμε, έχουμε και ένα ε, φιλικό προ το χρήστη ιντερνετικό εργαλείο που σα επιτρέπει να βρείτε μόνο σα τις πληροφορίες που χρειάζεστε είτε για χώρες είτε για αγορές. Φερρυπίν, μπορείτε να δείτε πώς πώς βαθμολογείτε μια αγορά μεταξύ των 50 στη χώρα σας ή σε όλη την Ένωση. Να δείτε ποια είναι η βαθμολογία για τις πέντε συνιστώσεις στη δική σας χώρα ή στην Ένωση. Ή να βρείτε και όλα τα γραφήματα που σας έδειξα για κάθε χώρα. Με τη βαθμολογία ένα χώρα. Μια ιστοσελίδα που μπορεί να μπει, στην οποία μπορεί να μπει ο καθένας μέσω του, της ιστοσελίδας της ΣΑΝΚΟ. Επόμενη διαφάνεια. Πέρα από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής για την αγορά, έχουμε και διάφορους πίνακες ε, σε ό,τι αφορά το scoreboard. Ίσως να είναι λίγο δύσκολο να τους διαβάσετε, αλλά αφορούν τις τιμές. Οι τιμές ασφαλώς ε, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για το καταναλωτή βασικός παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση. Στην ενιαία αγορά η απόκληση που υπάρχει, οι αποκλήσει στις τιμές στα διάφορα κράτη-μέλη, το οποίο, οι οποίε δεν εξηγούνται από την καταναλωτική δύναμη, από το κόστος, αποτελούν μια καλή ένδειξη της, του κατακαιρματισμού της αγοράς. Και γι' αυτό λοιπόν εξετάζουμε και αυτή τη διάσταση. Αυτό που δείχνει σε στον οριζόντιο άξονα η διαφάνεια αυτή είναι τις διαφορές ε, σε τιμή υπηρεσιών και προϊόντων σε διάφορες χώρες. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορές ε, στις τιμές που συνάδουν με την καταναλωτική δύναμη του καταναλωτή. Όσο πιο ψηλά είναι μια υπηρεσία και ένα αγαθό, όσο τόσο πιο πολλές διαφορές υπάρχουν στην καταναλωτική δύναμη. Και αντίστροφα, τα αγαθά που είναι κάτω από τον άξονα Χ Γι' αυτά ισχύει το αντίθετο. Είναι οι υπηρεσίε αυτές τα αγαθά πιο φτηνά σε χώρες όπου οι καταναλωτές είναι σχετικά πλούσιοι. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν. Αυτό ισχύει για παράδειγμα για κάποια αυτοκίνητα, για καύσιμα για αυτοκίνητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τιμές χωρίς τη φορολογία. Στην επόμενη διαφάνεια τώρα. τα αποτελέσματα τα οποία σας ε, έδειξα και τα οποία συνόψισα, γιατί υπάρχουν πολλά περισσότερα, ήταν από την ε, προηγούμενη έρευνα και προγραμματίζεται η διεξαγωγή μιας νέας έρευνας, 24 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει και πάλι 51 αγορές, αγορές θα εξεταστούν και πάλι και στην παρούσα φάση προσθέσαμε άλλο ένα ζήτημα, ένα θέμα ανταγωνισμού. Ρωτάμε λοιπόν τους καταναλωτές να μας πούνε σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10 εάν θεωρούν ότι υπάρχουν διαφορετικοί ε, έμποροι προμηθευτές από τους οποίους μπορεί να διαλέξει. Δεν έχουμε τα αποτελέσματα ακόμα όλα για, το αυτό, για την καινούργια αυτή έρευνα, αλλά συνολικά φαίνεται ότι οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί κάπως για τους καταναλωτές και βλέπουμε επίσης ότι γενικά οι καταναλωτές θεωρούν και κατατάσσουν τον ανταγωνισμό σε πιο υψηλές βαθμίδες από ό,τι άλλους δείκτες. Δηλαδή είναι πιο ευχαριστημένοι σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό από ό,τι είναι σε θέματα αξιοπιστίας, για παράδειγμα. Στην επόμενη διαφάνεια θα ήθελα να πω δύο λόγια και σε ό,τι αφορά τους καταναλωτικούς όρους στο σχετικό scoreboard των πίνακα αποτελεσμάτων που δημοσιεύεται την Άνοιξη. Εξετάζεται η ενσωμάτωση στην ε, λιανική εσωτερική αγορά. Κοιτάμε ε, διασυνοριακές πτυχές, ηλεκτρονικό εμπόριο και για παράδειγμα εξετάζουμε κατά πόσον εμπιστεύονται τις διασυνοριακές συναλλαγές οι καταναλωτές, κατά πόσον θα αγόραζαν κάτι σε μια άλλη γλώσσα, κατά πόσον και τι θεωρούν ως εμπόδιο στις διασυνοριακές συναλλαγές, τι τους ανησυχεί. Και έχουμε επίσης και κάποιες πληροφορίες για τα παράπονα που εκφράζονται σε ό,τι αφορά διασυνοριακές ε, συναλλαγές. Και πρόκειται πάντα για ενστάσεις οι οποίες ε, υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο διασυνοριακών συναλλαγών. Και βλέπουμε ότι περίπου το 1 τρίτο εξ αυτών αφορά τον τομέα των μεταφορών. Τονίζω ότι πρόκειται πάντα για διασυνοριακές συναλλαγές. Η δεύτερη πτυχή στην οποία εστιαζόμαστε είναι το καταναλωτικό περιβάλλον στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την προστασία του καταναλωτή και την εφαρμογή του σχετικού, της σχετικής νομοθεσίας. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε προέρχονται από το Ευρωβαρόμετρο σε ό,τι αφορά έρευνες και μεταξύ των καταναλωτών αλλά και μεταξύ των ε, εμπόρων. Και έχουμε καταρτήσει λοιπόν σχετικούς πίνακες με τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες, για παράδειγμα, ελέγχου εφαρμογής ε, σε ό,τι αφορά την, καταναλωτική, την προστασία του καταναλωτή, αλλά και την προστασία, την ασφάλεια των προϊόντων. Εδώ βλέπετε ένα πίνακα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μπορεί να γνωρίζετε τα αποτελέσματα αυτά, γιατί ε, έχει δημοσιευτεί σε πολλές άλλες γενικές διευθύνσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται. Είναι το πιο δημοφιλής τρόπος ε, διασυνοριακών συναλλαγών. Όλοι οι άλλοι τρόποι παρουσιάζουν πτώση. Αλλά βλέπετε ότι αυτό δεν ισχύει ιδιαίτερα για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Ισχύει κυρίως για το εγχώριο ηλεκτρονικό εμπόριο. Γιατί είναι πιο πολλά τα πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων που προσφέρεται. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε το μερίδιο των εγχώριων και των διασνοριακών συναλλαγών μέσω ίντερνετ. Και βλέπετε βασικά πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πολύ αναπτυγμένες σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Υπάρχουν επίσης και κάποιες άλλες χώρες, λογικά οι πιο μικρές χώρες, όπου το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πιο αναπτυγμένο όπως η Μάλτα, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, αλλά και η Κύπρος και η ε, Αυστρία, γιατί είναι πιο χαμηλέ τιμέ, πιο μεγάλη ποικιλία σε κάποια γειτονική χώρα ενδεχομένω. Και στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε τους όρους που επικρατούν στα κράτη-μέλη. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο σχετικό ε, δείκτη, ο οποίο καταμετρά κάποιες συγκεκριμένους παράγοντες, όπως για παράδειγμα η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στις αρχές, ε, η άσκηση και η χρήση, η συχνότητα χρήσης ένωμων μέσων. Όλοι αυτοί οι μεμονωμένοι λοιπόν δείκτες αποτυπώνονται στον κατάλογο αποτελεσμάτων σε ξεχωριστά φύλλα ανακράτος μέλος και εδώ βλέπετε λοιπόν το συνοπτικό κατάλογο. Και βλέπετε λοιπόν πάλι στον πίνακα αυτό πόσο διαφορετική είναι η όρη σε κάθε κράτος μέλος σε πόσο διαφορετική κατάσταση βρίσκονται οι καταναλωτέ σε κάθε χώρα. Στον επόμενο πίνακα βλέπετε λοιπόν ότι αποτυπώνεται η εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Και αυτό αφορά τρία ζητήματα, τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς, κατά πόσο εμπιστεύεται ο καταναλωτή ε, τις δημόσιες αρχές για να προστατεύσουν τα δικαιώματά του ως καταναλωτή. Κατά πόσο εμπιστεύεται τους εμπόρους, και το τρίτο ερώτημα, κατά πόσο θεωρεί ο καταναλωτής ότι προστατεύεται επαρκώς από τα εφιστάμενα μέτρα. Και βλέπετε λοιπόν πολύ διαφορετικοί οι όροι που επικρατούν άμα, στις διάφορες χώρες. Σε κάποιες χώρες, με κορυφαίο το Ηνωμένο Βασίλειο, 4 στους 5 καταναλωτές ε, θεωρούν ότι προστατεύονται παρκώς. Σε άλλες χώρες λιγότερο από το 1 τρίτο θεωρεί ότι είναι επαρκή η προστασία της οποία απολαμβάνει. Μεγάλες διαφορέ και εδώ. Στην επόμενη διαφάνεια. Εν συντομία. Φυσικά δεν μας ενδιαφέρει μόνο να παράγουμε ωραία αποτελέσματα. Όχι, κάτι θέλουμε να συμβεί. Θέλουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα αποτελέσματα. Άρα, τι κάνουμε συνομιλούμε πολύ με τα κρατημέλη και τα ενθαρρύνουμε να επικεντρώσουν τις προτεραιότητες τους στις αγορές εκείνες οι οποίες σημειώνουν κακό αποτέλεσμα σε εθνικό επίπεδο και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να θέσουν προτεραιότητες βάσει των αποτελεσμάτων. Επίσης, συνομιλούμε και με εκπροσώπους των επιχειρήσεων και τους καλούμε για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα και φυσικά αποτελώς στόχος είναι να βελτιωθεί η απόδοση ή τουλάχιστον η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Γιατί πολύ συχνά βλέπουμε ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν πάρα πολύ καλές πρακτικές για την προστασία των καταναλωτών και ότι ίσως να υπάρχει τρόπος να μεταφερθούν αυτές οι πρακτικές και σε άλλα κράτη. Επίσης, συνεργαστήκαμε με όλα τα όργανα ενστάσεων για να σε όλα τα κρατημέλη. Και καταλήξαμε σε κάποιες συστάσεις. Από του χρόνου, λοιπόν, θα υπάρχουν σχετικά στοιχεία συγκρίσιμα από κρατο μέλο σε κράτο μέλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν μπει στην διαδικασία ο καταναλωτή να υποβάλει ένσταση όχι μόνο στον έμπορο, αλλά και σε ένα τρίτο σώμα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικά κάποιο πρόβλημα στην αγορά. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Και τέλος, συνεργαζόμαστε και με την Eurostat και με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες, γιατί θέλουμε πιο πολλές τιμές σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες για να υπάρχει καλύτερη σύγκριση. Όπως είπα στην αρχή, διεξάγονται και έρευνες για τις αγορές. Τέσσερις ε, σχετικές έρευνες έχουμε ολοκληρώσει και εργαζόμαστε στην παρούσα φάση επί άλλων τεσσάρων. Και συχνά λοιπόν ε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι αμοιβέ είναι πολύ αδιαφανείς και προσπαθούμε λοιπόν σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές αμοιβέ, τις τραπεζικές, ε, τραπεζικά τέλη, να καταλήξουμε σε πιο διαφανή αποτελέσματα. Επίσης, ε, εξετάσαμε τέσσερις έρευνες σε ό,τι αφορά ...της εταιρείας ηλεκτροδότησης. Διεξήγαμε και μία έρευνα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες λιανικής πώλησης και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι πάντα εύκολη η σύγκριση. Οι άλλες έρευνες συνεχίζονται ακόμα και θα ολοκληρωθούν ε, σύντομα σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα σταματήσω. Κοιτάξτε αν θέλετε τον πίνακα των αποτελεσμάτων που έχουμε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα μας και στο dashboard. Και εγώ θα χαρώ, και εγώ και οι συνάδελφοί μου, να σα ε, διαφωτίσω με περαιτέρω πληροφορίες, τι οποίε ενδεχομένω να θέλετε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις ομιλητές έχω στον κατάλογο μου τώρα. Πρώτη η κυρία Γιάλα Σέντερ, μετά η κυρία Μάισερ, η Φώστερ, Λίχτενμπεργκερ, Μπιλμπάου. Η κυρία Γιάλα Σέντερ πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτον, να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την παρουσίαση αυτού, αυτής της ε, ενδιαφέρουσας ανάλυσης και των νέων προτάσεων ε, που κάνει για μελέτη για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα μιλήσω για την σχέση με τις μεταφορές και ιδίω την σχέση με την πληροφορική. Θα ήθελα λοιπόν να προβλέπει, δεν προβλέπεται, αλλά θα ήθελα να ασχοληθεί και ένα πιλωτικό σχέδιο για την δυνατότητα ε, πολυμεσικών κρατήσεων και σε υπερεθνικό επίπεδο. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, μπορείτε πέραν αυτών που μας δείξετε να μας πείτε τα εμπόδια που μπορεί να τύχουν, π.χ. ότι όταν έχεις περισσότερο του ενός ε, αεροσκάφη μπορεί να ανήκουν σε άλλες εταιρείε. Τι γίνεται, το δικαίωμα να κλείνει κανείς θέση σε τρένο που περνάει τα σύνορα. Ε, μετά, τι σκέφτεται για τις συνθήκες απαιτήσεων ή καταγγελίες. Δηλαδή όταν κάνεις μια, αυτή, μια υπερεθνική ε, αγορά, ξέρω εγώ, κράτηση στη Γερμανία για ισπανικά τρένα, υπάρχουν πάντα το προ, τα προβλήματα με τις προϋποθέσεις για να ζητήσεις για να κάνεις καταγγελία που δημιουργούν προβλήματα στην αξιοπιστία των μέσων αυτών και στην εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς αυτό το εμπόριο μέσω ίντερνετ. Έχετε κάποια μελέτη για τις προθεσμίες επίλυσης των καταγγελιών. Επίσης, μια εταιρεία που τη γνωρίζουμε όλοι και που συνεχώς υπάρχουν καταγγελίες, η Ryanair. Σκέφτηκε η Επιτροπή κάτι δημιουργικό, ούτω ώστε όπως οι καταναλωτές ελεύθερα μέσω blog ή Twitter να περιγράφουν τις ταλαιπωρίες που με την Α ή Β εταιρεία, με τη Ryanair ειδικότερα, γιατί αυτή έχει δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα. Έχει κάποια φόρμουλα, κάποια σκέψη για να χρησιμοποιήσει την, ε, τα blog αυτά για να καταγράφει δημόσια την, ε, το που μπορείς να κάνεις ε, καταγγελία. Γιατί ξέρετε με τη Ryanair ψάχνεις από εδώ, ψάχνεις από εκεί να βρεις κάποιον να, ε, να γράψεις κάτι και τελικά το βρίσκεις σου απαντάνε «Α, ξέρετε, δεν λήφθηκε». Μπορούμε λοιπόν με μια απλού, απλή φόρμουλα τύπου ε, name and shame να μειώσουμε τις, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Κύριε Μάισνερ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Δεν θα τα χρειαστώ τα τρία λεπτά. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ως Επιτροπή Μεταφορών θέλουμε περισσότερη κινητικότητα συνολικά για τις αγορές. Και αυτό είναι ένα βαρόμετρο του καταναλωτή, από τη σκοπιά του. Να δει δηλαδή τι χρειάζεται για να πάνε τα προϊόντα το α στο β. Και υπάρχει όμως και βαρόμετρο των παραγωγών για να δούμε τη σημασία των μεταφορών και για αυτούς. Επίσης ε, σκεφτόμουν γιατί ήταν τόσο χαμηλά στην κατάταξη οι σιδηρόδρομοι, ενώ είναι σημαντική για τους καταναλωτές, αν δούμε όλη την αγορά συνολικά. Τρίτον, τώρα έχουμε μία επισκόπηση και της δημοσκόπησης που κάνατε. Εσείς έχετε να μας δώσετε κάποιο δικό σας tip, Κάτι που δηλαδή που πρέπει ως Επιτροπή Τουρισμού και Μεταφορών να το προσέξουμε περισσότερα, εκτός από τα γενικά συμπεράσματα. Κάτι που να είναι για μας ας πούμε πολύ σημαντικό, γιατί εμείς θέλουμε να δράσουμε θετικά για τους καταναλωτές με αυτά που κάνουμε. Ε, μπορεί να υπάρχουν δηλαδή κάποια διαφωτιστικά στοιχεία που θα μπορούσατε εσείς να μας δώσετε. Η κυρία Φόρστερ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Κομισιόν για το έγγραφο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά ένα από, μια από τις πρώτες παρατηρήσεις, ερωτήσεις μου, είναι ότι λέτε συνέχεια εμείς, εμείς το ένα, εμείς το άλλο, εμείς ε, ρωτήσαμε την κοινή γνώμη. Ποιοι είναι αυτοί, είναι η γενική διεύθυνσή σας, είναι άνθρωποι ας πούμε που κάθονται και σηκώνουν ένα τηλέφωνο, κάθονται σε ένα τηλέφωνο και τηλεφωνούν ε, στην κοινή γνώμη ή είναι κάποιοι εθνικοί φορείς, γιατί υπάρχει και ένα ειδικό καλής πίστεως ε, περιοδικό στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο εξετάζει τέτοια θέματα και δεν είναι κυβερνητικό. Επίσης, μιλάτε για 500 ανθρώπους. 500 δεν είναι και μεγάλος αριθμός ε, για να εξεταστεί ένα συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι υποκειμενικές οι ερωτήσεις και δεν λέω να μην εξετάσουμε τα καταναλωτικά θέματα, αλλά είναι τόσο ευρύ το θέμα και τόσο περίπλοκο και φαίνεται να τίθενται τόσο διαφορετικά θέματα και καλύπτεται, πάτε να καλύψετε τόσα πολλά που δεν ξέρω ακριβώς τη σημασία. Και ποια ερώτηση, ας πούμε, περιμένετε, ε, ε, αν ταξιδέψετε με τρένο, με ρώτησαν πρόσφατα. Ε, ναι, είπα. Καλό το ταξίδι, ναι. Υπάρχουν κάποια παράπονα σε σχέση με αυτό, ναι. Γιατί πριν από δύο χρόνια που πήγα... δηλαδή είναι και παλιές οι πληροφορίες καμιά φορά. Ποιος αποφασίζει τι ερωτήσεις θα τεθούν. Υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση στα κράτη-μέλη. Αυτά είναι τα ερωτηματικά. Δεν λέω να μην μαζεύουμε πληροφορίες, βεβαίως χρειάζεται. Αλλά μιλάμε για το κόστος, ας πούμε, και για την Κομισιόν και για τους ε, καταναλωτές, τους ε, φορολογούμενους. Πόσο λοιπόν, στοιχίζει ένα τέτοιο έγγραφο, μια τέτοια έρευνα. Και ποιος το διαβάζει, ποιος είναι ο αποδέκτης, εγώ, η κοινή γνώμη. Δηλαδή, πού στοχεύει αυτή η έρευνα, ποιοι είναι οι τελικοί αποδέκτες. Και αν ένα κράτος μέλος δεν θέλει να συντονιστεί, ας πούμε, με τους φορείς του, τι θα κάνετε. Βλέπω ότι τα αλκοολούχα ποτά είχαν καλά αποτελέσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά εντάξει, τι να πούμε. Βεβαίω πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται σε ορισμένου τομεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή η, αυτή προσέγγιση είναι περίπλοκη με πολλού τομεί. Αυτά που είπε η κυρία Γιάλα ε, Ζέντερ, πούμε, δεν είναι ανόητος ο κόσμος. Επιλέγουν. Εγώ δεν θα πω, ας πούμε, ε, όπως είπε η κυρία ε, Τσέντερ για τη Ryanair, ο κόσμος έχει επιχειρήματα για να συγκρίνει και να προτιμήσει 35 εκατομμύρια. Ε, πιστεύουν ότι είναι καλή η Ryanair. Ε, δεν είναι σκοπός ο δικός μας να πούμε τι θα κάνει η κοινή γνώμη, τι θα κάνει ο κόσμος. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως και θα τους ενημερώνουμε με τρόπο σωστό, αλλά Ίσως πρέπει να γίνεται με απλούστερο και σαφέστερο τρόπο αυτό. Αυτές είναι κάποιες ερωτήσεις προς την Κομισιόν από μένα. Ευχαριστώ. Η κυρία Λίχτενμπέργεν, τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Αν ε, προβάλλουμε το επιχείρημα και το κάνουμε να ισχύσει και στη Ryanair, μπορούμε πολλά να ε, δικαιολογήσουμε και μπορούμε να υποβαθμίσουμε λίγο το θέμα της προστασίας των καταναλωτών έτσι. Αν, δηλαδή, αν κάποιοι αγοράζουν κάποιο προϊόν και δεν παραπονιούνται γιατί είναι δύσκολο να γίνουν καταγγελίες, γιατί αυτό είναι το θέμα, επειδή είναι δύσκολο να ακολουθήσουν την οδό της καταγγελίας. Δεν σημαίνει αυτό ή σημαίνει, όπως λέτε εσείς, ότι είναι ευχαριστημένοι. Και αυτό ισχύει και για την Επιτροπή μας και τους κανόνες μας. Εμείς θα πρέπει να δούμε Πώς είναι αυτοί που απελπίζονται ενώ πάνε να κάνουν μια καταγγελία και δεν συνεχίζουν. Και λένε, α, πολύ περίπλοκη και περίπονη διαδικασία ή ε, νιώθουν ενοχικά συναισθήματα γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με την ε, καταγγελία. Αλλά που δεν είναι αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση του καταναλωτή. Ούτε σημαίνει ότι εμείς ε, είχαμε νομοθετήσει σωστά επειδή μόνο ιδιαίτερα ευφυείς οι ικανοί ε, άνθρωποι ή ε, ε, μορφωμένοι μπορούν να φτάσουν να καταγγείλουν κάτι. Και πάω τώρα στην ίδια την παρουσίαση. Ευχαριστώ για το φυλάδιο. Προσπάθησα να το διαβάσω, αλλά δεν τα κατάφερα γιατί δεν είχα μαζί μου το μεγεθυντικό μου φακό. Όταν μιλάμε για καταναλωτές, και εδώ είναι 7 τα σημεία, δεν τα διαβάζει κανείς δημιουργούνται εμπόδια απαράδεκτα για μένα και αυτό ισχύει και για την παρουσίαση γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω τι έλεγε ε, το κάθε, η κάθε διαφάνεια. Είχα και τον υπολογιστή για να παρακολουθώ ταυτόχρονα αλλά πραγματικά είναι υπερβολικό εδώ μιλάμε για δημοσίευση της Κομισιόν και μιλώ και εκ μέρους των αναπήρων. Αν χρειάζομαι μεγεθυντικό φακό για να διαβάσω τα αποτελέσματα, δεν κάνει. Ε, αυτά για τον τρόπο της δημοσίευσης. Τώρα, η συγκρισιμότητα είναι ένα μεγάλο θέμα σε, πολλά, σε πολλές ε, στατιστικές και γλωσσικές παραδόσεις. Αυτό είναι σαφές. Και οι ερωτήσεις της συναδέλφου Φόρστερ ήταν σωστές από ό,τι μπόρεσα να παρακολουθήσω. Γιατί ρώτησε πώς συλλέγονται αυτά τα στοιχεία με το τηλέφωνο, πώς. Το στατιστικό δείγμα των 500 δεν είναι προβληματικό, αλλά σας ρωτώ, είναι ένα δείγμα που ισχύει σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, θα είναι το ίδιο μεγάλο το δείγμα στη Γερμανία και τη Μάλτα. Γιατί για αυτή την περίπτωση έχω κάποια στατιστική ένσταση. Ή διαφοροποιείται ας πούμε τα δείγματα ανάλογα με τις χώρες. Και τέλος και πολύ σημαντικό, τι τύχη τα περιμένει αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Αυτό εδώ είναι ένα έργο το οποίο θα το αναγνώσω με το μεγεθυντικό μου φακό όπως σας είπα, αλλά φοβάμαι ότι όταν μένουμε πολύ στην επιφάνεια δεν βγαίνουν αποτελέσματα τα οποία αυτά μας ενδιαφέρουν σε τελευταία ανάλυση στην Επιτροπή Μεταφορών γιατί θα επηρεάσουν και το νομοθετικό μας έργο. Ευχαριστώ. Ε, τα τυπογραφικά, <laughs> τα τυπογραφικά στοιχεία της έρευνας ε, έχουν το ίδιο μέγεθος όπως οι όροι και οι προϋποθέσεις της Ryanair. Ο κύριος Αούτζιας, τρία λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την παρουσίαση της δημοσίευσης ε, που μας έγινε. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Νομίζω ωστόσο ότι πρέπει να υλοποιηθεί η βάση αναφοράς, διότι η στατιστική βάση δεν είναι συνεπής. Ένα κράτος μέλος που έχει 60-80 εκατομμύρια πολίτες, το να ρωτήσουμε σε ένα τέτοιο κράτος 500 άτομα, ε, είναι ένα γεγονός που στερείται οποιασδήποτε στατιστικής ε, σημασίας. Σε οποιοδήποτε κράτος θα, ήταν, ε, θα στερεί το στατιστική σημασία. Δεύτερον, καλό θα ήταν να διευκρινίσουμε, και ελπίζω να το βάλετε αυτό στο site, ο τύπος των ερωτήσεων που τίθενται και ποιες ερωτήσεις τίθενται. Εγώ λοιπόν δεν ρωτάω καλό καλύτερα να υπάρξει μεγαλύτερη πρωτοβουλία για να αυξηθεί ο ρυθμός των ε, ερωτωμένων, για να έχει πραγματικά σημασία η ερώτηση. Κύριε Μπιλμπάου, τρία λεπτά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Επιτροπή για την παρουσίαση. Πέραν των μεθοδολογικών ζητημάτων που αμφισβητήθηκε και θα ήθελα και εγώ να έχω περισσότερες γνώσεις για τα στοιχεία και τα ποσοστά και δεν το επαναλάβω τόσο πάνω. Θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή το εξή. Όντω έγινε μια ανάλυση κρατών με βάση την κατάστασή του. Αν δούμε ωστόσο ένα από τα ζητήματα που αξιολογήθηκαν, Φερρυπίν, λειτουργία του τρένου, του τραμ, διακοπές, περιλαμβάνουν διαστάσεις που σε πολλά κράτη της Ένωσης αποτελούν αρμοδιότητα των περιφερειών, όχι του κράτους. Θα ρωτούσα λοιπόν, η ανάλυση που κάνετε και δεν φαίνεται να το κάνετε, μπορεί στο μέλλον τουλάχιστον να προχωρήσει στο εσωτερικό των κρατών μελών την κατάσταση δηλαδή ανά περιφέρεια, διότι οι τομείς που σας ανέφερα, αν δούμε τι γίνεται μεταξύ των περιφερειών της Ιταλίας, της Ισπανίας ή του Βελγίου, θα δούμε ότι η ανάπτυξη των δικαιωμάτων καταναλωτή είναι παράμετρος ή ε, η λειτουργία του τρένου, του τραμ, του των ξενοδοχειακών δομών. Δεν είναι αρμοδιότητα, ο έλεγχος δεν είναι αρμοδιότητα του κράτους. Πέρα λοιπόν του ποσοστού των ε, ερωτώμενων θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για το οποίο γίνεται θα είχαμε πολύ πιο θετικά αποτελέσματα αν κάναμε ανάλυση αναπεριφέρεια και θα βλέπαμε ότι πολλές περιφερειέ ξεπερνούν τα κράτη σε καινοτομία, σε άλλους τομείς και στην άσκηση ακόμα και την επίλυση των διαφορών. Η Ευρώπη είναι αποκεντρωμένη. Καλό λοιπόν θα ήταν να είχαμε και μια πιο αποκεντρωμένη εικόνα της κατάστασης. Ο κύριος Γκρός, τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ δεν είχα πολύ χρόνο να το εξετάσω το κείμενο. Μπόρεσα να διαβάσω ωστόσο. Να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η εργασία, αλλά οι ερωτήσεις που τέθηκα αφορούν και το προφίλ των ερωτηθέντων. Ίσως θα ήταν ε, ενδιαφέρον να δούμε το προφίλ των ερωτηθέντων και κατά δεύτερον οι καταγγελίες που έχουν ε, γίνει είναι ενδιαφέρουσες. Δεν μας αναφέρεται και ο ρυθμός των ε, καταγγελιών. Λείπουν λοιπόν πληροφορίες και κατά τρίτον το ερώτημα του τι θα γίνει μετά. Και αυτό νομίζω ότι αφορά ιδιαίτερα την Επιτροπή Μεταφορών. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν και κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμπεράσματα για την Επιτροπή μας και ίσως να καταρτιστούν και βέλτιστες πρακτικές. Γιατί υπάρχουν λιγότερα προβλήματα στις μεταφορές σε κάποιες χώρες και τι οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση σε άλλες χώρες. Διαπιστώσαμε, για παράδειγμα, ότι μεταξύ Βελγίου και Γαλλίας πάνω από 40% των οχημάτων άλλασαν τον αριθμό των χιλιόμετρων τους ε, σε ό,τι αφορά μεταφορικά οχήματα και πλέον υπάρχει μια κάρτα η οποία μετρά αυτά τα χιλιόμετρα και έτσι το αντίστοιχο ποσοστό πλέον έχει μειωθεί σε 0,8%. Με πολύ απλά μέτρα λοιπόν μπορούμε να καταπολεμήσουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν απλού τρόπου που δεν θα κοστίζουν ίσω και καθόλου χρήματα, αλλά θα προστατεύουν τον καταναλωτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Τιλ, θα μπορούσατε να απαντήσετε εν συντομία τι ερωτήσεις που σα έθεσαν οι βουλευτέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Να προσπαθήσω ό,τι μπορώ να το απαντήσω. Καταρχήν, μια ερώτηση για διασυνοριακές καταγγελίες και αν υπάρχει κάτι που το ετοιμάζομαι για τις καταγγελίες μίλησε και άλλο μέλος. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους καταναλωτές. Αν κάτι δεν πάει καλά δηλαδή να αποζημιωθούν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αυτό αποτρέπει πολλούς από ε, διασυνοριακές ε, συναλλαγές. Το ξέρετε περισσότεροι ότι τώρα ετοιμάζουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για εναλλακτική επίλυση διαφορών. Παράλληλα με αυτή την πρωτοβουλία θα υπάρξει και μία δεύτερη που στοχεύει ειδικότερα επιγραμμικές online συναλλαγές. Οπότε σύντομα θα έχουμε μία πρόταση τουλάχιστον για να βεβαιωθούμε ότι οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε online επίλυση διαφορών και αυτό πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για να ε, επιλύνονται τα προβλήματά τους. Ευτυχώς, α, δυστυχώς δεν έχουμε πληροφορίες για τους, ε, κα, ε, κατασκευαστές, γιατί έγινε μια ερώτηση σχετική. Ε, ζητήσαμε τις απόψεις των καταναλωτών. Ήταν πολλές οι ερωτήσεις σε σχέση με τη μεθοδολογία της έρευνας. Όλες τις λεπτομέρειες και τις εξηγήσεις όλα τα στατιστικά δεδομένα ε, υπάρχουν στην έκθεση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα βασικότερα ερωτήματά σας. Δεν ε, πήραμε συνέντευξη από 500 μόνο. Είναι 500 επί 50 αγορές, επί 27 κράτη-μέλη. Είναι πολλοί οι καταναλωτές που ερωτήθηκαν, δεν ήταν μόνο 500. Και αυτό έγινε μέσα από έναν ανάδοχο, γιατί δεν το κάνουμε εμείς ε, ή άμεσα. Προσπαθήσαμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα δείγματα των καταναλωτών που έδωσαν συνέντευξη θα ήταν όσο αντιπροσωπευτικότερα γινόταν σε όλο τον πληθυσμό, σε όλα τα εθνικά κράτη-μέλη και πράγματι ε, κάναμε συνέντευξη σε 500 κράτη-μέλη αλλά μετά επανασταθμίστηκαν τα ε, στοιχεία, τα νούμερα. Οπότε τα αποτελέσματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατοπτρίζουν τον πραγματικό πληθυσμό. Ε, φροντίσαμε, υποβοηθούμε και από την ε, Eurostat, ώστε να είναι όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευτικά γινόταν τα αποτελέσματα. Θέλαμε να πάρουμε περισσότερες συνεντεύξεις, αλλά δεν γινόταν. Θα ήταν πολύ δαπανηρή η μελέτη. Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για το αν μπορούμε να κάνουμε ε, πρωτότυπη ανάλυση. Αυτό ε, είναι πολύ θεμητό που ρωτάτε, αλλά Α, όχι πρωτότυπη, περιφερειακή, regional ε, ανάλυση να κάνουμε, αλλά με βάση τα δεδομένα και τη δομή τους δεν γινόταν προς το παρόν. Άλλοι μπορούν να το κάνουν αργότερα. Τώρα, για επιμέρους δράσεις και τι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχω όλες τις απαντήσεις εδώ. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Ανέφερα κανένα δυο, μιλάμε ε, με τα κράτη-μέλη για τα ζητήματα αυτά. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι συνάδελφοί μου που ήταν υπεύθυνοι για το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών ε, άρχισαν διάλογο με την ε, Lease Europe που ενοικιάζουν αυτοκίνητα και διευκρινίζεται η πληροφόρηση σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούν οι εταιρείε ενοικίασης αυτοκινήτων και θέλουν να κάνουν κι άλλο ένα βήμα. Όχι μόνο να είναι βέβαιοι ότι θα ενημερώνονται σαφέστερα οι καταναλωτές, αλλά θα εξετάσουν μαζί με τις επιχειρήσεις περισσότερο τα προβλήματα τα οποία αναφέρουν οι καταναλωτές στα κέντρα καταναλωτών και οι επιχειρήσεις ε, υποσχέθηκαν να ασχοληθούν με αυτά. Ήδη έχει γίνει αυτό. Αυτή είναι μία από τις δράσεις που ε, έχουμε, θα ακολουθήσουν και υπάρχουν ήδη και πολλές άλλες και ελπίζω και εσείς να ενθαρρύνετε τέτοιου είδους δράσεις από την πλευρά σας. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μας πιέζει ο χρόνος, είμαστε όμως πολύ ευγνώμονες που κάνατε την παρουσίαση απαντήσατε και στα μέλη. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα ακολουθήσει η συνεδρίαση των συντονιστών και οι υπόλοιποι θα έρθουν για να συνεχίσουμε ε, στις 9 με τις κάρτες ε, ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ακολουθήσει η συνεδρίαση των συντονιστών.